είναι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εξάλληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους. Η Επίτροπος Κρέτσου είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε το θέμα αυτό στην ημερησία την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Όπως ξέρετε το θέμα αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή. Και φυσικά δεν μπορούμε να ανεχθούμε ή να δεχθούμε οποιαδήποτε μορφή βίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό εξ αρχής. Ωστόσο, τα θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας δεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης αλλά των κρατών μελών. Η έμφυλη βία παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των θυμάτων και αποτελεί έκφραση της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η, η βία κατά των ε, γυναικών, μεταξύ των οποίων η σεξουαλική βία και παρενόχληση, είναι απαράδεκτη. Ανεξάρτητα από το background των δραστών. Όλοι πρέπει να σέβονται το νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η Ένωση. Η σεξουαλική βία δεν είναι νέο έγκλημα. Σε μια έρευνα της ΦΡΑ αποδεικνύεται ότι οι μισές γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αντιμετωπίσει σεξουαλική παρενόχληση. Πάνω από μία στις δέκα γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι είναι θύμα σεξουαλικής βίας μία στις 20 έχει υποστεί βιασμό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι δρόμοι μας, οι πλατείες, οι σταθμοί είναι ασφαλείς για γυναίκες και κοπέλες. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες δεν θα φοβούνται να αναφέρουν στην αστυνομία ή αλλού την σεξουαλική παρενόχληση ή βία σαν να πρόκειται για μια κλοπή και να διώκονται και να καταδικάζονται οι δράστες. Τα γεγονότα στην Γερμανία την τελευταία νύχτα του 2015 έδωσαν έμφαση στις ειδικέ διαστάσεις των σεξουαλικών επιθέσεων. Καλωσορίζουμε τα μέτρα που υιοθέτησε η Γερμανία ε, με ενίσχυση του, των ρυθμίσεων του ποινικού της κώδικα. Ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή σχετικών εμπειριών μεταξύ των Υπουργών Δικαιοσύνης. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας ε, και της οικιακής βίας κατά των γυναικών, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης όπως αποκαλείται, θέτει δεσμευτικούς κανόνες και πρότυπα σε διεθνές επίπεδο καθώ τα συμβαλώμενα μέρη πρέπει να καλούν να προστατεύσουν τι γυναίκε και τα κορίτσια από κάθε μορφή βία, μεταξύ των οποίων και τη σεξουαλική. Η Επιτροπή ε, εξετάζει και βρίσκεται σε εξελιγμένο στάδιο μία ε, πρόταση για μια σύμβαση πρώτο ε, για προσχώρηση στη σύμβαση αυτή της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ε, νομικά μέτρα για την υποστήριξη των γυναικών αυτών. Καταρχάς, ένα πρόβλημα είναι ότι, ότι ακόμα λίγες γυναίκες αναφέρονται στις αρχές για, τέτοια, για τέτοιες παραβιάσεις. Η οδηγία για την ε, ενίσχυση των θυμάτων ε, μπορεί να βοηθήσει την αύξηση των καταγγελιών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν το δικαίωμα για τα δικαιώματα των θυμάτων που επιτρέπει σε ε, θύματα δικημάτων και τις οικογένειές τους, υπηρεσίε μετάφρασης, προστασίας και υποστήριξης κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της δίκης. Οι τελικά χαρακτηριστικά της έμφυλης βίας υπογραμμίζονται στο πλαίσιο αυτό πρέπει οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη ειδικών, να υιοθετηθούν ειδικά μέτρα για την προστασία των ε, γυναικών κατά τη διάρκεια των, της δίκης, ενώ η Επιτροπή παρακολουθεί και θα παρακολουθεί την υλοποίηση της οδηγίας. Ξέρουμε ότι μόνο η νομοθεσία δεν αρκεί. Για το λόγο αυτό χρηματοδοτούμε έργα που επιτρέπουν να υπάρξει ε, πραγματικός αντίκτυπος στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών σε ό,τι αφορά την, ε, το να απολάβουν τα δικαιώματα της ισότητας. Έχουμε διαθέσιμα πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ για διεθνικά project ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων βίας και άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα για διεθνικά έργα καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε βαθιά δεσμευμένοι στο να πετύχουμε την ισότητα των φίλων. Οι προσπάθειες καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης πολιτικής μας για την ισότητα των φύλων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα επόμενα έτη θα λάβουμε μια σειρά δράσεων για τη βελτίωση της ισότητας μεταξύ των φίλων και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ευχαριστώ για την συζήτηση αυτό και θέλω να σας μεταβιβάσω το μήνυμα της συναδέλφου κυρίας Γιούροβα που δεν μπορούσε να είναι παρούσα εδώ σήμερα λόγω άλλων υποχρεώσεων που έχει εκτός Στρασβούργου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ενημερώνω το σώμα ότι σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες το Συμβούλιο δεν θα συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Ο πρώτος ομιλητής είναι η κυρία Χολμάιερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα γεγονότα της κολονίας την ε, βραδιά της πρωτοχρονιάς έχουν φέρει στο προσκήνιο τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών και έχουν προσδώσει μια νέα διάσταση στο θέμα αυτό και έχουν φέρει το θέμα στην επικαιρότητα. Υπήρξαν πολλές ε, πολλά βαριά αδικήματα στην περίπτωση αυτή με τράστες ε, ορισμένους προερχόμενους από το Μαρόκο και την Αλγερία που έκαναν σοβαρές παρενοχλήσεις. Αλλά φυσικά τα ίδια πράγματα πρέπει να ισχύουν και για αυτούς οι οποίοι δεν είναι μετανάστες και δεν προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική παρά όλα αυτά κάνουν τα ίδια και προβαίνουν σε σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική βία κατά των γυναικών. Κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο λοιπόν για τη Γερμανία να υπάρξει ποινικό κολασμός αυτών των ε, αδικημάτων και επομένως όπω ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υπάρξει η αλλαγή αυτή της νομοθεσίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να είναι σαφές ότι να μην είναι υποχρεωμένες οι γυναίκες να αποδείξουν ότι υπήρξε βία εναντίον τους και μόνο τότε να θεωρείται ότι υπήρξε αδικοπραξία. Κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες για τις γυναίκες. Επίσης όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι απογυμνωμένες από το δίκαιο. Ανεξάρτητα από την εθνικότητα του δράστη δεν πρέπει να υπάρχει ατιμορρεσία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες να μην τρομοκρατούνται <clears throat> και να μην επίσης να υποχρεώνονται να έχουν τους άντρες σε απόσταση, να μην φοράνε ποτέ μίνι φούστες κτλ. Να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες πρέπει να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων ελευθερίας που <clears throat> ε, πρέπει να απολαμβάνουν σε μια δημοκρατία και όχι σε ένα ε, Κράτο ολοκληρωτικό, όπου πολλές φορές η βία κατά των γυναικών θεωρείται αποδεκτή. Η κυρία Αρένα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Ευρώπη μία γυναίκα στις τρει ήταν ή είναι ή θα γίνει θύμα βίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ειναι η θα γινει θυμα βιας στι περισσοτερες περιπτωσει η βια ε, προέρχεται από ένα φίλο, από το σύζυγο, από φίλο της ε, οικογένεια όχι κατά ανάγκη ε, μετανάστη. 13.000 ε, γυναίκες το 2014. Το 2014 δεν είχαμε τη μεταναστική κρίση. Η Δία στην Ευρώπη δεν περίμενε τους μετανάστες για να πλήξει. Για μας, τους σοσιαλιστές, όλες οι γυναίκες θύματα βία θα πρέπει να τύχουν υπεράσπιση και όλοι οι δράστε να τιμωρηθούν, όποια και είναι η προέλευσή του, η τάξη του η θρησκεία του. Αυτό που έγινε στην κολονία είναι αξιολείπητο, αξιοθρύνητο. Θα πρέπει να εντοπίσουμε τους δράστες και να τους τιμωρήσουμε. Δεν ε, το μπορούμε να το κάνουμε όμως με ρατσιστική προσέγγιση, ε, ούτε στον δημόσιο χώρο, ούτε στον ιδιωτικό χώρο. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε μία ουσιαστική προσέγγιση, μία μέθοδο για να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, τις ε, κλασικές ιδέες ε, ότι ο άντρας είναι ο κύριος και η γυναίκα είναι το θύμα. Ο άντρας ο δυνατός, η γυναίκα αδύνατη, ε, ο άντρας ενεργητικός, η γυναίκα παθητική. Ας δούμε τις, ε, δήμωση, τις διαφημίσεις στην Ευρώπη για να δείτε πόσο αυτά τα στερεότυπα είναι εγγεγραμμένα στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Αυτή η συζήτηση δείχνει ακόμα μια φορά ότι το συνέστημα σκοτώνει τη λογική. Κάνω έκθεση στη λογική για να κάνω μια δουλειά μακροπρόθεσμη, όπω μια στρατηγική Φερρυπίν που ψηφίσαμε σήμερα το πρωί υπέρ τη ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Ευχαριστώ. Κυρία Βυσνιέσκα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν τεράστιος αριθμός επιθέσεων στις πόλεις της Ευρώπης κατά γυναικών. Δείγμα του ότι η πολυπολιτισμικότητα απέτυχε. Δεν είναι τυχαίο το ότι δεν αντέδρασε η γερμανική αστυνομία την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Κάποιοι είπαν ότι το προκάλεσαν τα θύματα, ότι τα θύματα προκάλεσαν τις επιθέσεις με τον ντύσιμό τους μας υποχρεώνουν στο σπίτι μας να προσαρμοζόμαστε στους κανόνες άλλων χωρών. Ο κύριος Τίμερμανς είπε για την κολονία ότι υπήρξε πρόβλημα δημόσιας τάξης που δεν σχετίζεται με τη μεταναστευτική κρίση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πόσο, πόσο καιρό περιμένει η Ένωση για να σταματήσει να θεωρεί ότι καλύτερη είναι μεταναστευτική πολιτική από την ασφάλεια των γυναικών της. Ξέρετε τι γίνεται στα κέντρα προσφύγων. Πότε θα σταματήσουμε να μιλάμε και να θέσουμε πέρας στη βία κατά των γυναικών. Πότε θα αναλάβουμε δράση του ώστε οι γυναίκες στην Ευρώπη να αισθάνονται ασφαλείς. Με, με τρομάζει πόσο τυφλή μπορεί να είναι κάποιοι στις νέες μορφές βίας και των γυναικών σε σχέση με την ε, μεταναστευτική κρίση. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ εντυπωσιάζομαι από την ξαφνική ανάδυση κύματος φεμινισμού σε όλη την Ευρώπη. Βλέπω να βλέπω γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του Eurostat 25% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι μία κοπέλα που φοράει φουστά, τα ζητάει. Προκαλεί προβλήματα. Είναι πολύ απλό γιατί και οι επιθέσεις της κολονίας χρησιμοποιήθηκαν ρατσιστικά και λαϊκιστικά για να δημιουργήσουν το, το μίσος κατά των μεταναστών. Δεν έπαιξε ρόλο εκεί καθόλου το πρόβλημα της παρενόχλησης γυναικών. Τι γίνεται όμως το Oktoberfest, τις γιορτές του Οκτωβρίου στο Μόναχο με τις γυναίκες οι οποίες επίσης χουφτώνονται εκεί. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να υπάρξει η υποστήριξη στις γυναίκες που δεν είναι οπορτουνιστικού χαρακτήρα. Τα γεγονότα λοιπόν της κολονίας δεν πρέπει να θεωρηθούν προβλήματα ενσωμάτωσης των μεταναστών πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση για τον ρόλο των γυναικών. Όχι μόνο στα πλαίσια τη συζήτηση για τη μετανάστευση, αλλά μέσα στην ευρωπαϊκή κοινωνία γενικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια αντιμετώπιση που δεν εξαρτάται από πού προέρχονται αυτές οι γυναίκες ή ποιοι επιτίθενται εναντίον τους. Χρειαζόμαστε μια ενιαία αντιμετώπιση και να υπάρξει αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Προφανώς υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πιθανότητα για, ένα, για μια εγκληματική ενέργεια κατά των γυναικών δεν εξαρτάται από αυτές τις πολιτιστικές διαφορές. Πρέπει να έχουμε θετικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε και την, το κύμα των προσφύγων και να τους ενσωματώσουμε στις κοινωνίες μας. Εάν λοιπόν δει κανείς όσο λίγοι είναι οι πρόσφυγες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, θα καταλάβετε ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από την κυρία Λεμπέσιου. Είστε έτοιμοι να απαντήσετε. Λεμπέσιου. Frau Melina, Sie haben gesagt, ähm, dass äh, Sie haben gesagt, dass 25 äh, Prozent äh, oder dass Schülerinnen aufgefordert werden, keine Minimum. Είπε ότι στα σχολεία πολλές φορές ε, ζητούν από τα κορίτσια να μην φοράνε μινιφούστες, ότι 25% των, Γερμανών, των ερωτημένων, ερωτηθέντων θεωρούν ότι μια κοπέλα φοράει μινιφούστα προκαλεί με την ενέργειά τους και λέτε ότι αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τους πρόσφυγες και αναφερθήκατε ότι στην Oktoberfest υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Δεν υπάρχει με 5 εκατομμύρια οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα τέτοιο είδος επιθέσεων όπως αυτές που αναφέρθηκαν στην ε, ε, κολονία. Τι πιστεύετε για όλα αυτά. Αυτές ε, οι πληροφορίες που μας λέτε θα πρέπει να σας πω ότι είναι εσφαλμένες. Αυτό που εγώ παρέθεσα ήταν έρευνα της Eurostat και δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία είπατε εσείς, ή μάλλον ισχυριστήκατε εσείς. Επίσης ξέρουμε ότι η βία εις βάρος των γυναικών εκδηλώνεται ανεξάρτητος του ποιος είναι ο υπέτειος και όταν εκδηλώνεται πρέπει να αντιμετωπίζεται. Σε αυτό δεν έχω καμία επιφύλαξη. Αλλά δεν θα παρασυρθώ στον οπουρτινισμό των καιροσκοπικών φεμινίστριων για να πω ότι θα ακολουθήσω τα δικά σας επιχειρήματα. Το Björk. Πρόεδρε, είναι ουσιώδους χαρακτήρα αυτή η συζήτηση. Όταν ε, τα κορίτσια βλέπουν ότι μπορεί στο δημόσιο χώρο να βρίσκονται σε δυσμενή θέση, να βρεθούν σε δυσκολίες, σε σχολεία, ε, συναυλίες, ε, στο δρόμο, ότι μπορεί να υπάρχει μια σεξιστική προοπτική, ότι μπορεί να πέσουν θύματα παρενόχλησης γυναίκες ή κορίτσια. Δέχονται και σεξιστικές απειλές συχνά από άντρες. Και εμένα μου έχει συμβεί να δεχθώ από λευκούς Ευρωπαίους άντρες. Η σεξιστική απειλή εις βάρος των γυναικών είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο και σεξιστικες απειλες συχνα απο αντρες και μενα μου εχει συμβει να δεχθω απο λευκους ευρωπαιους αντρες η σεξιστικη απειλη εις βαρος των γυναικων ειναι ενα πανευρωπαικο φαινομενο και πρεπει να την καταπολεμήσουμε ως τέτοιο. Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ε, πηγαίνει ανεμπόδιστη να καταγγείλει στην αστυνομία. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για μια πιο φεμινιστική Ευρώπη. Δεν ανεχόμαστε πια να υφαρπάζει τα κορμιά μας η άκρα δεξιά για να προβάλλει ρατσιστικά επιχειρήματα. Το γυναικείο σώμα είναι θέμα ελευθερίας, είναι θέμα αυτοδιάθεσης, είναι θέμα δικαιώματος στην άμβλωση, είναι θέμα πάνω απ' όλα ελευθερίας. Σήμερα σας βλέπω εδώ να μιλάτε, αλλά την τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει για τα θέματα της ε, ε, ε χειραφέτησης των γυναικών δεν ήσασταν παρόντες. Τώρα μόνο για να πείτε ότι μας απειλούν οι πρόσφυγες σας εδώ. Πρέπει κάθε μέρα να γίνεται αυτός ο αγώνας για τις γυναίκες και για την ε, προστασία τους. Ευχαριστώ. Κυρία Μπιόρκ, έχετε μια μπλε κάρτα της κυρία Βυσνιέσκα που διέχεστε. 30 δεύτερα. Ευχαριστώ. Ε, αξιότιμη κυρία, δεν θεωρείτε ότι το, το επιχείρημά σας αποκλείει κάποιους, γιατί αυτά που είπατε ε, και οι ορισμοί που δώσατε για τους ε, ευρωβουλευτές δεξιών πτέρυγων νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή σε μία ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πραγματικά η δική σας ρητορική είναι ρητορική μίσους. Και αν ε, είχατε ανοίξει τα μάτια σας θα βλέπατε ότι και χθε καθόμουν στην ίδια θέση. Μπορώ να διαπιστώσω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ και συζητούμε τα θέματα αυτά, πάντοτε τα ζητάσουμε υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, υπέρ τη αυτοδιάθεση. Εσεί, είτε πρόκειται για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, είτε πρόκειται για τα δικαιώματα των παιδιών, των γυναικών, να καθορίσουν μόνε του τη ζωή του, πάντα καταψηφίζετε, πάντα τάσεστε κατά σε οτιδήποτε είχαμε να συζητήσουμε στο πεδίο αυτό εδώ στην Ευρώπη. Προφανώ δεν σα ενδιαφέρει να περασπιστείτε τι γυναίκε, αλλά θέλετε να διαδώσετε το ρατσιστικό σα μήνυμα. Σας ευχαριστώ κυρία Άρεντ και εκ μέρους των Πρασίνων Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η σεξουαλική βία και παρενόχληση είτε κατηδίαν είτε στους δημοσίους χώρους δεν θα πρέπει να είναι θέμα ταμπού. Η σεξου... Η πρόσθεση σεξουαλικού χαρακτήρα στη βία είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αναλαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν εξαλειφθεί αυτή η βία, ποτέ δεν θα πραγματώσουμε την ουσιαστική ισότητα που προβλέπεται και από τις συνθήκες. Θα πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά στην ισότητα. Και γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίζουμε τις, ε, τις εκστρατείες ε, αφύπνισης της συνείδησης. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση γυναικών και κοριτσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς το καλύτερο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν ακόμη σε ό,τι αφορά το σεξουαλικό χαρακτήρα που έχει η η παρενόχληση. Και φυσικά θα πρέπει να μιλήσουμε για τη φαλοκρατία, για την πατριαρχική κοινωνία και χειραφετημένες ελεύθερες γυναίκες που ε, επιλέγουν ελεύθερα για τη ζωή και το κορμί τους απειλούν τη φαλοκρατική ανδροκρατούμενη κοινωνία. Θα πρέπει να τα πούμε αυτά με ξεκάθαρο τρόπο. Όπου σε όποιον τομέα και αν μιλούμε. Και δεν θα πρέπει φυσικά να θεωρούμε από διαπομπέους τράγους συγκεκριμένες ομάδες, ε, ούτε να ε, υποθάλπουμε ρατσιστικές, ε, ρατσιστικά μίση. Νομίζω πριν από λίγο καιρό ε, με κατηγορούσαν για φεμινιστικές βλακίες και τώρα με απειλούν για, γιατί προσπαθώ να προάγω τη θέση των γυναικών. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να, κανείς να σφετερίζεται την ελευθερία μου και το κορμί μου, το κορμί των γυναικών για να προαγάγει ε, πολιτικούς σκοπούς αν θέλουμε ισότητα για όλους θα πρέπει να σκάψουμε πιο βαθιά, να βρούμε τις ε, ρίζες του κακού και να χτυπήσουμε τα αίτια του. Και δεν θα πρέπει να ενδίδουμε σε υπεραπλουστευτικές συζητήσεις, ε, ρατσιστικές ε, και τελείως περιτές. Η κυρία Μάρκοτ Πάρκερ από την Ευρώπη των Ελευθεριών και Δημοκρατιών για τρία λεπτά. Ναι, νομίζω ότι Καλό να καθόμαστε εδώ και να λέμε ότι θέλουμε ανοιχτέ πόρτε, αλλά πραγματικά ο κόσμο υποφέρει και είναι παράξενο που η Κομισιόν δεν αποδέχεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αυτή τη ε, προσφυγική κρίση και των επιθέσεων στην κολονία. Πράγματι, με αποκάλεσε ένα εργατικό ε, ρατσίστρια όταν μίλησα για αυτέ τι επιθέσει. Αν ήμουν η μητέρα σα, η κόρη σα, η φίλη σα, δεν θα δεχόσασταν ακόμα ότι δεν συνέβη τίποτα. Αυτό συνέβη όταν ανοίγουμε την πόρτα σε άλλες χώρες και πολιτισμούς που μεταχείριζονται τις γυναίκες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Μετέχουμε τις ε, καλυμμένες συνέργειες αστυνομίες και των άλλων αρχών και δεν λένε ακριβώς την αστυνομία, η αστυνομία τι γίνεται επειδή ακριβώς θα μπορούσε να ωφελήσει κάποια πολιτικά κόμματα και το να γίνονται αυτές οι, το να υπάρχουν αυτές οι δράσεις είναι ατυχές. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε την ασφάλειά μας, αλλά λόγω ακριβώς της πολιτικής ε, ορθότητας ε, δεν κάνουμε το σωστό. Τι γίνεται όταν θα έχουμε αυτούς τους ανθρώπους με διαβατήρια με εθνικότητες από αυτές τις χώρες. Θα έρχονται λοιπόν σε αυτές τις χώρες μας χωρίς να ελέγχεται το μητρό τους. Το 2015 είχαμε 100.000 παρόμους πρόσφυγες που ήρθαν στην, που ήθελαν να πούν στον Ανωμένο Βασίλειο. Αυτό δείχνει ακριβώ το μέγεθο τη κρίσεω. Και βλέπουμε ότι πάνω από 10.000 παιδιά προσφύγων έχουν εξαφανιστεί. Τα παιδιά λοιπόν αυτά και οι νέοι έχουν υποχρεωθεί σε σεξουαλική εκμετάλλευση από κάποια αποδίκτυα. Υπόθηκε μάλιστα ότι πολύ συχνά πολλά από αυτά τα παιδιά θα εμπλακούν σε αυτά τα δίκτυα εκμετάλλευση. και Αυτά φαινόμενα έχουμε λοιπόν από την Μεσόγειο και όλες αυτές οι απειλές για τις γυναίκες, για τα παιδιά, αφορούν ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν μια ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για να διευρύνει το νόημα της συνθήκης της Γενεβής για αυτούς που φεύγουν από συγκρούσεις και έχουν με εκατομμύρια που φτάνουν στην Ευρώπη το 2015, πολλοί χρειάζεται να προσφύγουν σε εγκληματικέ οργανώσεις για να φτάνουν να φτάσουν εδώ. Και η ελεύθερη διακίνηση τους επιτρέπει να έρθουν εδώ. Δεν υπάρχουν έλεγχοι μητρώου και η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί μια τεράστια απειλή ασφάλειας, όπως είδαμε και από τις θερμοκρατικές συνεργασίες στο Παρίσι. Και γραφούν λοιπόν ελεύθερα στην Ευρώπη, επιτίθενται σε ελεύθερους δημόσιους χώρους χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θέτει τι γυναίκε σε άμεσο κίνδυνο και νομίζω ότι αποτελεί την πηγή αυτή τη κρίση. Η ασφάλεια λοιπόν των γυναικών και άλλων αυτών θυμάτων μας υποχρεώνει να ελέγξουμε τα σύνορά μα και να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πάρκερ, μια μπλε κάρτα. Την κυρία Ρέντκε. Θέλετε να τη δεχθείτε. Όχι. Δεν σας ακούω. Όχι. Όχι, μάλιστα, δεν τη δέχεται. Η κυρία Βίκη ένα λεπτό. Η Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, είμαι εξοργισμένη ε, κατά της ευρωπαϊκής ελίτ που όλο μιλά και λέει ωραία λόγια για την ασφάλεια αλλά δεν λέει τίποτα για τον κίνδυνο εξισλαμισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί απειλή για τις γυναίκες. Το είδαμε στην Κολονία, στη Φραγκφούρτη και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι γυναίκες γίνονται θύματα βιασμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης γιατί λαμβάνει η χώρα ένας χωρα ένα ένα μια σεξουαλική τζιχάντ. Μερικοί ε, το θεωρούν ως ζήτημα μετανάστευσης, αλλά είναι ζήτημα δημόσιας τάξης. Πώς ε, τολμάτε να χρησιμοποιείτε τόσο ε, σκανδαλώδη επιχειρηματολογία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σέγγεν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο χώρος Σέγγεν, αυτό διευκολύνει τη σεξουαλική τσιχάτ που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη και ανοίγει τις πύλες στον Ισλαμικό, στην Ισλαμική βαρβαρότητα. Θα πρέπει να αποισλαμίσουμε τις χώρες μας. Κύριος Η άλλη Σφάρτσερ. Αγωνίστρα για τα δικαιώματα των γυναικών, έχει περιγράψει αυτή τη βία ως το υποπροϊόν μιας αποτυχημένης, ποτέ σωστά σχεδιασμένης ε, κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αποτελεί το απάβγασμα της μυσαλλοδοξίας πέρας της παραθέσεως. Μια πολιτική λοιπόν των ε, ανοιχτών συνόρων και της διαλλακτικότητας ή της ανοχής, κακώς νοουμένης ανοχής που επέδειξε άλλωστε και η κυρία Μέρκελ, όπου είπε ότι θα δεχθεί πρόσφυγες και θέτει εκτός λειτουργίας το Δουβλίνο και το Σέγγεν. Στις ευρωπαϊκές πόλεις με πρώτη την κολονία η βία που εκδηλώθηκε εις βάρος των γυναικών προκύπτει όχι λόγω ε, αποτυχίας δράσης της αστυνομίας αλλά γιατί ξαφνικά απειδείχθη πως δεν μπόρεσαν να κατακρύψουν να καταπνίξουν τις ειδήσει οι στατιστικές. Μάλιστα καταγγέλθηκαν ε, τα γεγονότα ως ε, κίτρινος τύπος. Αυτά δεν έχουν καμία θέση στην Ευρώπη και πάνω απ' όλα σε κανένα εθνικό κράτος. Ευχαριστώ. Η κυρία Κωνσταντς Λουκρύπ, δύο λεπτά. Πρόεδρε. προχωρημένη ώρα που συζητάμε σήμερα και το έχουμε συζητήσει εδώ και ασχολούμαστε με θέματα δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητας ανδρών και γυναικών και για να συζητήσουμε για νέα επεισόδια βίας εις βάρος των γυναικών και σεξουαλικής παρενόχλησης τους. Ε, δεν το πράττουμε επειδή το έχουμε συνήθιο ή κάποιο είδους τελετουργικό μια φορά το χρόνο, παρότι θα έπρεπε ίσως να αφιερώσουμε μια φορά το χρόνο επί τη ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας ε, για ε, να μιλήσουμε για την ε, βία εις βάρος των γυναικών, για να τονίσουμε κάποια στοιχεία κτλ. Αλλά γιατί υπήρξαν γεγονότα, γεγονότα κατάφορα τα οποία προξένησαν κλειδονισμού σε όλη τη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη και εδώ μιλάμε για μαζικές παρενοχλήσεις σεξουαλικές ε, εις βάρος γυναικών στην Κολονία και άλλες πόλεις Γερμανίας της την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ένα πρωτοφανές γεγονός, μια βία μαζική και άκρος ε, μαζική και βία η κατάληψη του δημόσιου χώρου από ομάδα ανδρών που εκδηλώθηκε άξαφνα η βία εις βάρος των γυναικών δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε εθνότητα, ούτε θρησκεία, ούτε χρώμα δέρματος, η φαλοκρατία, ο ανδρικός σοβινισμός, η βία εις βάρος των γυναικών, η ενδοοικογενειακή βία δεν ανήκουν σε καμία εθνοτική ή άλλη ομάδα και αυτό το καταγγέλουμε πολύ συχνά στα έδρανα εδώ του Κοινοβουλίου και κυρίως όταν ε, ε, Έχουμε την επέτειο της, ε, του αγώνα, της ημέρας για τον αγώνα κατά της βίας παρός των γυναικών τον Νοέμβριο. Καταγγέλουμε τα γεγονότα αυτά παγίως. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε και να κλείσουμε τα μάτια, δεν μπορούμε να αποστρέψουμε το βλέμμα ή να αρνηθούμε την πραγματικότητα. Δεν έχουν συμβεί σε τέτοια διαστάσει και ένταση τέτοια γεγονότα στο παρελθόν και μια γαλίδα και αριστερή φιλόσοφος μας καλεί να σταθούμε στο πλευρό. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Μικέλα Τσουφρίτα, δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα γεγονότα της κολονίας σοβαρότατα θα πρέπει να διχτούν με τη μέγιστη ευθυρότητα. Δεν θα πρέπει όμως να χρησιμεύσουν για να δώσουν χώρο σε μια διαμάχη λαϊκιστική που θα καταστρέψει την Ευρώπη. Η καταδίκη θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Γνωρίζοντα όμω ότι είχαμε να κάνουμε μια πραγματική τρομοκρατική ενέργεια που είχε μελετηθεί μέχρι τελευταία λεπτομερία για να αποσταθεροποιηθεί η όλο και πιο ευαίσθητη ισορροπία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να γενικοποιήσουμε αδιάκριτα και να στρέψουμε το δάχτυλο κατά όλων των προσφύγων. Εκείνη η επίθεση, εκείνο το βράδυ, είχε διοργανωθεί με τρόπο ημιστρατιωτικό, προβλέποντας ακριβώς και τις επιπτώσεις. Μία επιχείρηση λοιπόν όχλησης τόσο μεγάλη δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μία χειρονομία κατά των γυναικών. Είναι μια χειρονομία πρόκλησης κατά όλης της κοινωνίας μας, του πολιτισμού μας, της ελευθερίας μας. Το να εντοπίσουμε και να δείξουμε ξένους μετανάστες και πρόσφυγες δεν θα βοηθήσει στο να αποτρέψουμε τη βία κατά των γυναικών. Αυτά τα επεισόδια σοκάρισαν όλο τον κόσμο. Όμως ακόμα οι γυναίκες της πόλης μας παραμένουν θύματα όχλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι δυστυχώς ακόμα είναι ριζωμένη μια νοοτροπία και ένας πολιτισμός της γυναίκας ως αντικείμενο. Χρειάζονται λοιπόν σοβαρότατα και αυστηρότατα μέτρα καταδικαστικά, αλλά κυρίως η νοοτροπία της κατάχρησης και της αυθαιρεσίας που θα έπρεπε να καταπολεμηθεί. Καταρχάς με την εκπαίδευση για τον σεβασμό του ατόμου που βρίσκεται στην βάση για τον σεβασμό των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζουγκέρη και ένα λεπτό και τριάντα δεύτερα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λάθος είναι όταν διαφωνεί κανείς με κάποιον να καταγγέλει τον συναδελφό του ως ρατσιστή. Κυρία Κρέτσου, η κολονία πια έχει μετατραπεί σε σύνθημα για την βία εις βάρος των γυναικών, αποτυχία των αστυνομικών αρχών, κατά εγκληματικών οργανώσεων. Αυτό μας το ζούμε σε όλη την Ευρώπη. Όλοι θέλουμε να σταματήσει η σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος των γυναικών και όχι μόνο στο δημόσιο χώρο. Μια γυναίκα στις τρεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από πολύ νωρίς, δηλαδή 62 εκατομμύρια γυναίκες. Κάθε 68 ε, λεπτά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας μια γυναίκα στη Γερμανία. Πρέπει να, πέσει, να έρθει ένα τέλος λοιπόν σε αυτήν την υπόθεση. Σεξουαλική παρενόχληση και επιθέσεις στην παραμονή της πρωτοχρονιάς ε, έδωσαν πλέον, ε, έκρουσαν το κόδωνα του κινδύνου για την ανάληψη μέτρων που, έχει, που χρειάζεται να έχουν ληφθεί εδώ και καιρό. Πρέπει η συζήτηση λοιπόν να γίνει αντικειμενικά, πρέπει να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα με αποδεικτικά στοιχεία να διωχθούν οι ε, δράστες αλλά βέβαια πρέπει να υπάρξει και μια δράση αξιολόγησης των σεξουαλικών αυτών αδικημάτων ε, ανάλογα με την ένωμη τάξη κάθε κράτους που είναι διαφορετική η σεξουαλική παρενόχληση βάρος γυναίκας παραδείγματι θεωρείται μόνο έργο εξύβριση ενώ θα μπορούσε να είναι άσκηση βίας. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε. Κύριε και έχει περάσει ο χρόνος σας. Έχει περάσει ο χρόνος σας. Κύριε Γκέρικε αντιμετωπίζω όλους τους ε, ισότιμα και έχει περάσει ο χρόνος σας. Η κυρία Μπέατρης Μπεσέρα Παστερετσιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δράστε των παρενοχλήσεων και οι βιαστέ είναι εγκληματίες και, οι εγκληματίε ε, πρέπει να διώκονται, να δικάζονται και να τιμωρούνται. Όποιοι και αν είναι, όπου και αν βρίσκονται και από όπου και αν προέρχονται. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Το θέμα είναι πώ θα δράσουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Ολλανδική Προεδρία για την επικείμενη κύρωση τη σύμβαση ε, Σύμβασης της το πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο που καλύπτει σφαιρικά το θέμα τη βία κατά των γυναικών. Ερωτώ λοιπόν το Συμβούλιο θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του κλήρωση τη ε, σύμβαση αυτή και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση φέτο, όπω ήδη επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστόματο Επιτρόπου Γιώροβα. Έχουμε την πολυτέλεια μήπω ε, να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό το νομικό εργαλείο. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν είναι αποτελεσματική η οδηγία για τα θύματα των ε, εγκλημάτων που θεσπίσαμε το 2012. Θα γίνει κάποια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή στην Ένωμη μεταξύ των κρατών μελών για να δούμε αν εφαρμόζεται μια και έχει λήξει ήδη προθεσμία μετάθεσής της. Ευχαριστώ κυρία Κορνίλια Άνστη για ένα μισή λεπτό. Όταν ε, άκουσα τα όσα είχαν συμβεί στην κολονία μου κόπηκε η αναπνοή γιατί έλαμβανε νέες διαστάσεις πλέον ε, η φαλοκρατική παρενόχληση σφαρός των γυναικών. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά δεν πρέπει και να επιτρέψουμε να αξιοποιηθεί η συζήτηση αυτή για, όλου, για άλλους σκοπούς, για τους ναζί, για τους ρατσιστές, για αυτούς που θέλουν να ξεφορτωθούν με λίγα λόγια τους πρόσφυγες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ε, παραγνώριση της αξιοπρέπειας της γυναίκας με προσβολή της, πατριο... της ε, αξιοπρέπειας της γυναίκας που προέρχεται από πατριαρχικές δομές και θεωρήσεις. Έτσι πρέπει να περιγράψουμε το πρόβλημα. Δεν είναι απλώς διατάραξη της τάξης η παρενόχληση σεξουαλικής βάρος γυναίκας. Δεν πρέπει να, έχει, να φοβάται πλέον μια γυναίκα να πάει στο δικαστήριο και να καταγγείλει αυτόν που της έχει επιτεθεί. Δεν μπορεί η αστυνομία να αποστρέφει το βλέμμα όταν βλέπει τέτοιου είδους επιθέσεις βάρος των γυναικών, παρενόχληση μέχρι και βιασμό. Πρέπει να φροντίσουμε πλέον οι βίες βάρος των γυναικών να ε, εκφραστεί ως ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλες τις σωστές του διαστάσεις και όχι ως, ένα, ε, ως μια παρεπίπτουσα συνέπεια, συνέπεια μιας άλλης επιλογής. Πρέπει να ε, υπάρξουν προγράμματα υποχρεωτικά ε, για τη διαπαιδαγώγηση στα θέματα της αξιοπρέπειας των γυναικών σε όλα τα κράτη-μέλη, για την ισότιμη μεταχείριση, για το δικαίωμα στη ζωή, για τη δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει κανένα, καμία πραγματική ελευθερία χωρίς το, αν δεν τεθεί τέρμα σε αυτό το πρόβλημα για τις γυναίκες. Ευχαριστώ. Ορτασούν ένα λεπτό. ευχαριστώ. Τα γεγονότα της κολονίας, όπως οποιοδήποτε γεγονός βίας κατά γυναικών, είναι ατυχή και θα πρέπει να διωχτούν. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ εδώ σε αυτό που είπατε κάποιοι από εσά, το να μιλήσουμε για τους πρόσφυγες. Γιατί αυτό το φαινόμενο βίας κατά γυναικών είναι γενικό και όχι μόνο ευρωπαϊκό. Κάποιοι προαλήσαντες είπαν ότι υπάρχει μια έκθεση από το Ινστιτούτο κατά τη ε, βία των γυναικών που λέει ότι των τρίτων γυναικών έχουν υποστεί ένα είδο ε, βία στην Ισπανία ακόμα περισσότερο. Είχαν πολλά θύματα, πέρσι 54, 16 μέχρι τώρα από την αρχή του έτου. Οπότε αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε γενικά και μια καλή. Ένα καλό μάθημα σήμερα μετά από αυτή τη συζήτηση είναι ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό το είδος καταστάσεων και αυτό φαινόμενο γενικά στο σύνολό Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Επιτροπέ. Δεν γίνεται η συζήτηση αυτή να γίνεται τόσο αργά και ένα μήνα μετά τα γεγονότα. Στις γερμανικές πλατείες είχαμε ένα παιχνίδι διασμών δεν είναι μια υπόθεση δημοσιογράφων αυτό, αλλά η κατάληξη του και το συμπέρασμα του, της γερμανικής αστυνομίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα εγκληματικό δίκτυο ανδρών που διέσαν γυναίκες. Και εμείς το καταδικάζουμε. Από όπου και αν προέρχεται. Στην Αφρική, στην Ασία, στην Ευρώπη. Εγώ δεν θέλω να βλέπω να καταπατώνται τα δικαιώματα και ελευθερίες που έχουμε κατακτήσει εμείς οι γυναίκες. Η Κομισιόν θα πρέπει να αποδείξει συγκεκριμένα ότι θα αντιμετωπίσει και θα βάλει τέλος αυτή τη μάστιγα της βίας και να μην κρύβεται πίσω από αυτή την σιωπή της. Οι γυναίκες δεν χρειάζονται κουβέντες, αλλά δράση. Κυρία Κολονία, Ντίσελτορ, Στοκόλμη, Στουτγκάρτη, Ζηρίχη, Αμβούργο. Σε όλε αυτέ τι πόλει εκατοντάδε γυναίκε έπεσαν θύματα βιασμού ή σεξουαλική παρενόχληση χρήα μορφή από ορδέ ε, μεταναστών. Και παρόλα αυτά οι αρχές έμειναν ε, σιωπηλές. Βέβαια οι ε, φεμινιστικές οργανώσεις καταδίκασαν τις φαλοκρατικές αντροκρατούμενες κοινωνίες, ενώ αυτοί που ουσιαστικά και κατηγόρησαν τους ρατσιστές και τη Μαρίλε Πέν που έχησαν το ρατσιστικό τους μίσους εις βάρος των μεταναστών. Σας διαβεβαιώ ότι το Εθνικό Μέτωπο είναι το πιο φεμινιστικό του, του γαλλικού πολιτικού τοπίου, γιατί εμείς ταχθήκαμε κατά του, το φαινομένου αυτού. Επίσης στη Γαλλία κανένα σημαντικό πολιτικό κόμμα δεν είναι κατά του δικαιώματος των γυναικών σε άμβλωση. Το θέμα είναι ότι ο κίνδυνος για τις γυναίκες προέρχεται από μια ανεξέλεγκτη μετανάστευση και οι πατριώτες που εκπροσωπώ εγώ είναι η καλύτερη έπαρξη για την προστασία αυτών των γυναικών. Ευχαριστώ. Κυρία Καλπέλτσε, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στη συζήτηση αυτή, η οποία ε, αντιμετωπίζει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ταυτόχρονα όμως αισθάνομαι και βαθύτερη τη θλίψη. Γιατί φαίνεται πως πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ακόμη δεν μπορούμε να συζητήσουμε ανοιχτά και ελεύθερα. Ένα φαινόμενο το οποίο κάποτε φαινόταν απόμακρο, ο κίνδυνος μακρινός, φαίνεται τώρα να είναι πρώτον θυρό, να είναι μέσα στις κοινωνίες μας. Διπράχθησαν εγκλήματα εις βάρος γυναικών, νεαρών γυναικών και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και πρέπει να αντιδράσουμε κατά της βίας με πολιτική μηδενικής ανοχής. Πρέπει να σταματήσουμε να σιωπούμε, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε ανοιχτά. Πώς μπορεί η δήμαρχος να λέει ότι δεν μπορεί ε, ότι, ότι δεν πρέπει τα κορίτσια να φοράνε μίνι φούστες ή αρώματα στο δρόμο. Πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ανοιχτά. Αυτοί οι άνθρωποι δοκίμαζαν μέχρι που τους έπαιρνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στη χριστιανική κουλτούρα οι γυναίκες πάντα ήταν, ε, την χάναν ιδιαίτερου σεβασμού και δυστυχώς τώρα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Η κυρία Μούντι δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνώ με του αδελφού για την καταδίκη αυτών των επιθέσεων κατά των γυναικών στην Ευρώπη την παραμονή τη Πρωτοχρονιά. Παρ' όλα αυτά, η όχληση των γυναικών δεν άρχισε την 31η Δεκέμβρη 2015. Πράγματι, δύο μήνε νωρίτερα είχαμε τη γιορτή τη πύρα στο Μόναχο, όπου εκατοντάδε γυναίκε ανέφεραν σεξουαλικέ οχλήσει. Φαίνεται ότι δεν υπήρξε μεγάλη ανησυχία για εκείνε τι γυναίκε. Επίση, η Υπηρεσία Θεμελιδών Δικαιωμάτων αναφέρει ότι το 2014 μία στις τρεις γυναίκες ήταν αντικείμενο βίας. Οπότε η όχληση των γυναικών δεν είναι νέο φαινόμενο. Η βία και οι διακρίσεις στην Ευρώπη προηγούνται των γεγονότων της κολονίας και αλλού. Εγώ ήμουν ανέκαθεν κατά αυτών των δράσεων και των δραστών και είμαι περήφανη που και εγώ και οι συναδελφοί μου έχουμε υιοθετήσει συγκεκριμένα βήματα για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, παρόλα αυτά όσο το έκανα αυτό, ποτέ δεν είδα αυτούς που φώναζαν πολύ να μου συμπαρασταθούν για να πολεμήσουμε για τα δικαιώματα των γυναικών στο παρελθόν. Έχω λοιπόν αμφιβολίες για το UKIP και για το εθνικό μέτωπο της Γαλλίας την ξαφνική μετατροπή τους υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Υποψιάζομαι ότι επιθυμούν να υπάρχει φόβος και μίσος και όχι να προστατεύσουν τα θύματα. Αλλά ελπίζω να είμαι λάθος. Ελπίζω και εύχομαι το Ηνωμένο Βασίλειο να προσυπογράψει τη συνθήκη της ε, Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών των γυναικών. Ελπίζω Εν τω μεταξύ, ας προσπαθήσουμε να προωθήσουμε πολιτικέ που θα προστατεύουν τις γυναίκες από την εμπειρία αυτή της όχληση, ό,τι και να χρειαστεί να γίνει και ανεξαρτήτως δραστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μούντι, έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Γιούρεκ, τη δέχεστε. Όχι. Η κυρία Ουλρίκε Τρεμέσιους, ένα λεπτό και τριάντα δεύτερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα τα περιστατικά της κολονίας. Σε 200 πόλεις Γερμανίας είδαμε αντίστοιχε επιθέσεις. Είτε πρόκειτο για θόπευση, είτε πρόκειτο για ληστεία με σεξουαλική παρενόχληση, είτε πρόκειτο για βιασμούς. Φαίνεται ότι γεγονότα τέτοια έχουν μετατραπεί σε ορισμένε περιοχές σε καθημερινά φαινόμενα. Οι γυναίκες βλέπουν να αλλάζει η καθημερινή τους ζωή. Πρέπει να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους ε, και, αν, ε, και κινδυνεύουν να πέσουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους χωρίς να έχουν την ε, προστασία από κανέναν. Υπάρχουν δήμοι που σκοπεύουν από ό,τι φαίνεται να δημιουργήσουν στα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς ε, ζώνες αποκλειστικά για γυναίκες που θα τις σηματοδοτούν με ροζ χρώμα. Βλέπουμε, ροζ χρώμα. Βλέπουμε να μην αντιδράει η πολιτική ε, τάξη της Γερμανίας. Βλέπουμε οι αστυνομικέ αρχές να μην έχουν τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα μέτρα. Βλέπουμε να ε, φροντίζει η αστυνομία τους πρόσφυγες περισσότερο παρά τα θύματα αυτής της τόσο αποτυχημένης κοινωνικής ενσωμάτωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερώνουν και το Συμβούλιο της Ευρώπης την προηγούμενη εβδομάδα με ένα ψήφισμά του ε, προειδοποίησε και συνέστησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην περιορίζονται μόνο στο πολιτικό σορθό αλλά να μεταφέρουν αυτά κάθε αυτά τα γεγονότα. Πρέπει και εμείς να υποστηρίξουμε αυτές τις θέσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Μπαραντή, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τα επεισόδια παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας ε, οργανωμένου χαρακτήρα που έλαβαν ε, χώρα την περασμένη χρονιά σε πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, ούτε συνδέεται μόνο με την μεταναστευτική κρίση. Είναι απαράδεκτο να γίνεται κάτι τέτοιο βάρος των γυναικών. Το είδαμε την 1η Ιανουαρίου, αλλά θα αλλάξει η κατάσταση όταν καταλάβει ο κόσμο ότι είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά ει βάρο των γυναικών. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην ισότητα, γιατί η ανισότητα όχι μόνο θίγει τι γυναίκε, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ω διαρθρωτικό πρόβλημα, γιατί τέτοιο είναι. Τέτοιου είδου επιθέσει είναι ένα πολύ δυσάρεστο σταθερό στοιχείο πολλών ε, τομέων και συμπεριφορών. Και πολλές φορές ε, γίνονται συμπεριφορές ε, και ο βιασμός μερικές φορές και εργαλείο ε, πολέμου που κάνει τις γυναίκες θύματα. Και μάλιστα γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία, στην εξάλληψη των στερεοτύπων, μηδενική ανοχή εις των δραστών και η συμπερίληψη και των ανδρών στην προσπάθεια και σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι θα, θα βελτιώσουμε και την ένταξη. Ο κύριος Ζωάν Πιμέντα Λόπες, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα επεισόδια που καταγράφηκαν ε, στα τέλη του έτους στην Κολονία είναι πολύ σοβαρά. Οι σεξουαλικές επιθέσεις βάρος των γυναικών ε, και μάλιστα ο οργανωμένος ε, φαινομενικά χαρακτήρας τους δημιουργούν ένα πλαίσιο που χρήζει ε, πλήρη διαλεύκανση των πραγματικών περιστατικών ε, πέραν ε, της χειραγώγησης που προσπαθεί να κάνει άκρα δεξιά και της ρατσιστικής επιχειρηματολογίας που χαρακτήρισε μερικές φορές την ανάλυση τους. Μάλιστα, θα πρέπει να σταματήσουμε του εσφαλμένου συνειρμού και συνδέσμου μεταξύ τη προσφυγική ροή και των επεισόδιων τη κολονία. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τη συζήτηση στο βασικό και ουσιώδε πρόβλημα, τη σεξουαλική παρενόχληση και βία βάρο των γυναικών. Βία οποιασδήποτε μορφή ει βάρο των γυναικών. Για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, τη συμπεριφορά αυτή των ε, φυσικών αυτούργων και να βελτιώσουμε την ισότητα των δύο φύλων. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε απερίφραστα τα δικαιώματα των γυναικών, να επιβεβαιώσουμε την αξιοπρέπειά του και να προωθήσουμε ουσιαστικέ πολιτικέ ισότητα των δύο φύλων, κάτι που δυστυχώ ακόμη παραμελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σούρτη, Σεβαστία, ένα Αντίθετα με άλλου συντρόφου, εγώ θα μιλήσω για το θέμα που μα απασχολεί απόψε. Όπω είπε ο σύντροφο Φορτασούν, θα προωθήσετε επιτέλου μια οδηγία ευρωπαϊκή κατά τη βία ε, τη φυλετική, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Μιλάμε για βία κατά των γυναικών σε δημόσιου χώρου. Υπάρχουν όμω και φαινόμενα σε ειδικού χώρου. Και υπάρχει βία κατά των γυναικών, γιατί συνεχίζουμε αυτά τα τριπαρχικά κλισέ, τα οποία συγκρότησαν αυτή την ευρωπαϊκή κοινωνία. Κάποιοι συνάδελφοι κλείνουν τα μάτια και κατηγορούν τους ε, μετανάστες. Είδαμε τα στοιχεία. Μία στις τρεις Ευρωπαίες γυναίκες είναι θύμα βίας, όχι από πρόσφυγες. Αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι μια ευρωπαϊκή ντροπή, ένα όνειδος μένουν τιμώρητοι οι δράστες. Χρησιμοποιείται η γυναίκα με τρόπο τροπιαστικό στη διαφήμιση. Αυτό δημιουργεί στερεό, στερεότυπα ώστε ακριβώς να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η βία. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή θα κάνει κάτι για να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ένα Κυρία Πρόεδρε, πολλά συζητήθηκαν, πολλά υπόθηκαν για τα γεγονότα της κολονίας και, για άλλες, ε, και σε άλλες πόλεις. χρόνο βλέπουμε να ε, επεκτείνεται ο λαϊκιστικός ε, ρατσισμός στις χώρες μας. Πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λογικό. Γιατί πρόκειται για γυναίκες των διαφορετικών εθνοτικών προελεύσεων, θρησκευτικών ομάδων είτε όχι, είναι απαράδεκτο να πέφτουν θύματα τέτοια ε, βία. Ο καθένα ή κάθε μία πρέπει να αισθάνεται ασφαλή μέσα στι πόλει μα και πρέπει να καταστήλουμε με ε, αμήλικτο τρόπο αυτού που προσπαθούν να ε, αποκρύψουν την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει, και το λέω απερίφραστα αυτό, καμία δικαιολογία νοοτροπίας ή πολιτιστικής ε, προέλευσης για τα όσα συνέβησαν στην ε, κολονία ή για οτιδήποτε άλλη πράξη βίας. Όπως και να δίνεται κανείς, όπως και να είναι η εμφάνισή του, όποιον και να αγαπάει, όπως και να κυκλοφορεί στον δρόμο, έχει δικαίωμα να ζει ελεύθερος από φόβο και να κυκλοφορεί στους δρόμους. Αυτό είναι άλλωστε και ο πυρήνας των ευρωπαϊκών αξιών και πρέπει βεβαίως να εγγυόμεθα τα δικαιώματα των πάντων. Ταυτόχρονα θεμητό είναι να απαιτούμε οι θεμελιωδέστερες των αξιών να ε, τη προστασία στην Ήπειρο για οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε υποκείμενο τους. Ευχαριστώ πολύ. Post. Δύο λεπτά. Ο πατριαρχικός σοφινισμός βεβαίως συζητείται πλέον με αυτούς τους όρους. Η φαλοκρατία επιτέλους μπήκε στην ημερήσια διάταξη, θέλω να υπογραμμίσω. Όμως το φαινόμενο ούτε καινούριο είναι, ούτε εστιάζεται ή χαρακτηρίζει κάποια συγκεκριμένη εθνικότητα, εθνότητα, κοινωνική ομάδα ή προέλευση. Η βία των ανδρών εις βάρος των γυναικών έχει πανδημικό χαρακτήρα, είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει θύμα σεξουαλικής σωματικής βίας. Και πολύ, το, πολύ συχνά αυτή η βία εκδηλώνεται μέσα στην ίδια την οικογενειακή αιστεία της γυναίκας. Εδώ πρέπει να δώσουμε απαντήσεις λοιπόν. Δεν ναι, μπορεί μια γυναίκα να αισθάνεται ασφαλής μέσα στο ίδιο της το σπίτι ή στο δρόμο που θα κυκλοφορήσει. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στο οποίο πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει απαντήσεις. Πρέπει πλέον να δράξουμε το πρόβλημα και να δώσουμε απαντήσεις ανησυχητικό δεν είναι, το, δεν είναι η εθνοτική προέλευση των δραστών, αλλά το ότι δεν υπάρχει επαρκής προστασία. Δεν ήταν μεμονωμένα τα φαινόμενα και τα γεγονότα της κολονίας. Είναι πολύ συνηθισμένο από διαφορετικές εθνοτικές προελεύσεις ή κοινωνικές ε, τάξεις άνδρες να παρενοχλούν ε, σεξουαλικά οι γυναίκες. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να μην αφήσουμε να μετατεθεί η αιστεία του προβλήματος από ορισμένου εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Πρέπει τώρα να δώσουμε επιτέλους απαντήσεις στη Σουηδία. Είχαμε μια εκστρατεία η οποία οδήγησε στη συνέχεια ε, στο να, πάρουν, να κατέβουν στους δρόμους ρατσιστές για να επιτεθούν εις βάρος ε, ε, προσφύγων. Δεν ανήκουν αυτοί στη σουηδική κουλτούρα. Κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ και την καταδίκη των γεγονότων της κολονίας. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι ναι, είναι αλήθεια ότι δεν ανακάλυψαμε μόλις τώρα τη βία κατά των γυναικών και θα ήθελα να αναφέρω αυτό που έκανα πριν 40 χρόνια ως ε, φοιτήτρια δεκαετία του 70 είχαμε ένα κίνημα του να διεκδικήσουμε τη νύχτα και προσπαθούσαμε δηλαδή να επιτρέψουμε στις γυναίκες να βγουν το βράδυ ή τη νύχτα μόνες τους όπως επιθυμούσαν χωρίς όχληση μιλάω για τον Ηνωμένο Βασίλειο εδώ έτσι είναι λοιπόν απαραίτητο να δώσουμε, ήταν απαραίτητο τότε μάλλον να δώσουμε την δέουσα προσοχή και δεν μιλούσαμε τότε βέβαια για την Ισλαμοποίηση της Ευρώπης, δεν είχαμε να κάνουμε με πολιτιστικά ζητήματα, μιλούσαμε καθαρά για την Βρετανία. Και οι άντρε τότε δεν επέτρεπαν στις γυναίκες να συμπεριφερθούν φυσιολογικά. Και δυστυχώ βρισκόμαστε στην ίδια θέση ακόμα. Και ελπίζω το μάθημα της κολονίας να μας διδάξει ότι πρέπει να πάμε στα πραγματικά αίτια αυτού του φαινομένου και να αλλάξουμε πραγματικά τη ζωή για τις γυναίκες. Ελεονόρα Φορέντσε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω τα συμβάντα της κολονίας θα πρέπει να κρυθούν με βάση την αλληλεγγύη χωρίς υποσημειώσεις για τις γυναίκες που έχουν υποστεί αυτή τη βία. Νομίζω ότι η αλληλεγγύη με τις γυναίκες αποτελεί το σημείο κίνησης για οποιαδήποτε τοποθέτηση σχετικά με αυτό που συνέβη. Νομίζω ότι μια πραγματική πολιτική κατά της βίας των γυναικών, κατά της αντρικής βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να ξεκινάει από την διασφάλιση της πύρης, της πύρους ε, χειραφέτησης και νομίζω ότι η βία η αντρική θα πρέπει να καταπολεμηθεί η οποία είναι και ηλική αλλά και συμβολική. Οι γυναίκες χρησιμοποιούνται ως αντικείμενο όταν χρησιμοποιούνται και σε εκστρατείες ξενοφοβικές και ρατσιστικές. Όπως έλεγε η προελή σας ο συνάδελφος, εμείς δεν χρειαζόμαστε προστάτες, δεν χρειαζόμαστε αφεντικά ούτε στρατούς. Ευχαριστώ. Κύριος Μπούχνερ, ένα λεπτό. Σε μια ελεύθερη Ευρώπη πρέπει οι ελεύθερες γυναίκες και το βράδυ ελεύθερα και χωρίς φόβο να μπορούν να κυκλοφορούν. Αυτό δεν συμβαίνει πια στην Ευρώπη όμως και είναι, αποτελεί σκάνδαλο. Σε αυτό η πέτειο είναι σε μεγάλο βαθμό το υπερβολικά χαλαρό ποινικό δίκαιο το οποίο αντιμετωπίζει ως πτέσματα τα φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης βάρος γυναικών. Ταυτόχρονα έχουμε την προοπτική της υποδοχής ενός εκατομμυρίου πλέον πολιτών, ανδρών επιτοπλίστων. Κάθε χωρίο βέβαια έχει την αστυνομική του δύναμη, το αστυνομικό του τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές λοιπόν εν ώψη αυτών των εξελίξεων των δημογραφικών θα έπρεπε να είχαν ενισχυθεί, αλλά αντί να ενισχυθούν ε, έχουν ε, μειωθεί οι αστυνομικές δυνάμεις και γι' αυτό αντί να παραιτηθεί ο αρχηγό τη αστυνομία στην κολονία, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο υπουργό των εσωτερικών και πολλοί άλλοι υπουργοί μαζί με αυτόν. Ο κύριο Σφαίρ, ένα λεπτό και τριάντα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω κάτι για τον τίτλο ε, αυτής της συζήτησης, για το κεντρικό θέμα. Γιατί δεν ε, λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Πρόκειται για συγκεκριμένες εκδηλώσεις βίας σε συγκεκριμένο τόπο εις βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων. Γιατί μιλούμε εδώ για σεξουαλική βία εις βάρος των γυναικών σε δημόσιους χώρους και ούτω καθεξής. Σίγουρα είμαστε καλοπροαίρετοι και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφευθεί η επανάληψη τέτοιων φαινομένων, να μην έχουμε επεισόδια σαν αυτά της κολονίας και αλλού. Αλλά αυτά, αυτές οι εκδηλώσεις βίασης βάρος των γυναικών στην κολονία δεν ήταν κάτι τυχαίο. Ήταν πραγματική οργανωμένη επίθεση βάρους του συστήματός μας ε, και θα πρέπει να είμαστε άτεγκτοι, αμήλικτοι στο μήνυμά μας. Κανείς δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας. Κανείς δεν πρόκειται να μας αναγκάσει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και διαρωτώ για ποιο λόγο πολλές γυναίκες και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις αισιόπισαν. Δεν είπαν τίποτα, δεν σχολίασαν καθόλου τα επεισόδια αυτά. Προσπάθησαν μάλιστα να αποσπάσουν την προσοχή μας σε άλλα θέματα, στην ενδοοικογενειακή βία. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι χάσαμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε πραγματικά και ειλικρινά και σταράτα για αυτό που συνέβη. Η επόμενη ε, ομιλήτρια είναι η κυρία Τόμασιτς για ένα λεπτό. Η σεξουαλική παρενόχληση και η βία εις βάρος των γυναικών είναι απολύτως απαράδεκτη σε κάθε περίπτωση και θα πρέπει να τιμωρούνται αυστηρότατα. Φυσικά όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει στους τέσσερις στίχους ενός σπιτιού, μερικές φορές είναι αδύνατο να αντιδράσουμε και η κακοποίηση δεν βγαίνει στο φως. Αντίθετα, όταν αποφεύγουμε δρακόντια ακύρωση της, βίωσης, της βίας σε δημόσιους χώρους, είναι τελείως αδικαιολόγητο. Είμαστε μάρτυρες μιας αναδικής τάσης ε, της ε, δημόσιες κακοποίησεις των γυναικών στην Ευρώπη που είναι άμεση συνέπεια ελλειπούς ε, κοινωνικής ένταξης μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη από μη, πολιτισμικ... από μη ευρωπαϊκές πολιτισμικές σφαίρες. Δυστυχώς όμως μέχρι τα τελευταία επεισόδια της ε, Γερμανίας πολλοί έκαναν τα στραβά μάτια λόγω πολιτικής ορθότητας. Αυτό πάντως ε, δεν είναι πλέον δυνατό. Τέτοια αντιπολιτισμική συμπεριφορά είναι από τη σκοπιά του νόμου και της ηθικής απολύτως απαράδεκτη και θα πρέπει να εξαλειφθεί θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι ο νόμος ισχύει για όλους και για τους ε, μετανάστες και τους ε, ετούντες άσυλο και όσοι δεν είναι έτοιμοι να το δεχτούν αυτό δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στην Ευρώπη. Ο κύριος Στέφαν Εκ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, φυσικά καταδικάζω απερίφραστα τις ε, επιθέσεις της κολονίας και διερωτάται κανείς πώς μπορεί να προστατευτούν οι γυναίκες ε, κατά των σεξουαλικών αυτών επιθέσεων, γιατί πάνω από 30% των γυναικών στην ε, Γερμανία πέφτουν μέχρι τα 16 τους ε, θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βία. Δεν μπορούμε όμως να επιτρέψουμε η παραμονή της πρωτοχρονιάς στην κολονία να πέσουν στα χέρια των ακροδεξιών κομμάτων εδώ του Κοινοβουλίου για τη ρατσιστική τους προπαγάνδα και να ε, δημιουργήσουν συναισθήματα μίσους εις βάρος των προσφύγων, σαν να ήταν ο σεξισμός ή η σεξουαλική βία κάτι το πρωτοφανές στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί, επειδή προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική να θεωρούνται υπέτειοι αποκλειστικά και μόνο για αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να αγωνιστούμε κατά του, ρατσισμού, κατά του, ε, της φαλοκρατίας, κατά της ξενοφοβίας. Γιατί αλλιώς θα κάνουμε μεγάλο κακό στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Άννα Σαμπόρσκα. ένα λεπτό και τριάντα. Δεύτερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, μια από τις κύριες αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προστασία και ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου, άνδρα, γυναίκα, σύμπη, ζήτημα μόνο πολιτιστικής παράδοσης ε, στην Ευρώπη, είναι και ε, κανόνας της ένομης τάξης. Είναι Καταδικαστέ, λοιπόν κάθε τέτοια παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ιδιαίτερα όταν τα θύματα είναι γυναίκες. Δεν έχει σημασία αν ο δράστης της βίας είναι πολίτης ε, του εν λόγω κράτους, μετανάστης ή πρόσφυγας. Η σύμβαση της, γυναίκη, της Γενέβης επιτρέπει την απέλαση πρόσφυγα εφόσον έχει καταδικαστεί για ε, ποινικό αδίκημα. Πιστεύω ότι η αξιπρέπεια των γυναικών πρέπει να ταξινομηθεί στα, στις αξίες που η προσβολή τους χαρακτηρίζεται ως κακούργημα και μόνο έτσι μπορούμε να δούμε ένα τέρμα σε αυτές τις απειλές. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι οι μετανάστες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια. Καλό τις χώρες να τροποποιήσουν τη σχετική τους νομοθεσία με στόχο να προστατέψουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλων των πολιτών της Ευρώπης. Ευχαριστώ. γιουρέ και ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στην κολονία συνέβη κάτι φρικτό, αλλά δυστυχώς επαναλήθηκε και σε άλλες πόλεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, περίμενα μια σοβαρή συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά πραγματικά απογοητεύτηκα τα μάλα από αυτά που άκουσα στη συζήτηση. Η ταπείνωση των γυναικών είναι ένα γενικό φαινόμενο και αυτό που συνέβη στην Πολωνία δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Πολύ συχνά οι γυναίκες αποσιωπούν τέτοιες συμπεριφορές και τέτοια κακοποίηση. Οπότε στην, ε, στην Γερμανία το αποσιώπησε η αστυνομία. Αυτό συμβαίνει και όχι μόνο στη Γερμανία, έχει συμβεί και αλλού. Πρόκειται για θέματα γενικά. Αυτό όμως που θα πρέπει ε, να αναφέρουμε εμείς ε, είναι ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε τη συζήτησή μας στο εξή. Έχω ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει, στυλιτεύει τη συμπεριφορά της αστυνομίας που αποσιώπησε τέτοιου είδους εγκληματικές συμπεριφοράς. Ε, στυλιτεύει την αποσιώπηση για πολιτικούς λόγους ε, τέτοιων συμπεριφορών. Και μάλιστα θεωρεί ότι καταπατούνται αρχές ε, του άρθρου 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήθελα παρακαλώ να σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος ε, Μιγγέλ Ουρμπαν Κρέσπο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Το τέλο των επιθέσεων αυτών, το σεξουαλικό κατά των γυναικών, πρέπει να αποτελέσει μια απόλυτη προτεραιότητα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συζήτηση είναι κενή αν δεν μιλήσουμε για τα πραγματικά και βαθιά αίτια τη βία κατά των γυναικών. Α μην δείχνουμε κινησμό. Οι επιθέσει αυτέ δεν καθορίζονται από την εθνικότητα ή την οικονομική κατάσταση του δράστη, αλλά από, το, από τη φαλοκρατία που είναι ριζωμένη στην κοινωνία μας. Και κάτι άλλο, η άκρα δεξιά και η δεξιά, όπως βλέπουμε, προσπαθούν να στιγματίσουν τους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες για να προσπαθήσουν να κερδίσουν μία ούφτα ψήφους και παραβλέπουν τις καθημερινές σεξουαλικές επιθέσεις που γίνονται στα σύνορά μας, στο εσωτερικό των σύνορων μας, από Ευρωπαίους άντρες σε μια κοινωνία που θεωρείται πολιτισμένη. Οι γυναίκες λοιπόν ζουν υπό αυτό τον ζυγό. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε ώστε τα λόγια να μετατραπούν σε δράσεις για να αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει να τελειώνεται λέει Πρόεδρος. Τελείωσε. Κυρία Σόιτροβα, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δίνω αγώνα για την καταπολέμηση της βίας βάρος των γυναικών, όχι επειδή είμαι φεμινίστρια, αλλά γιατί η προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί προτεραιότητα των χριστιανοδημοκρατών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε δυστυχώς ότι η βία εις βάρος των γυναικών δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Όπως αναφέρθηκε ήδη, 30% των γυναικών αντιμετώπισαν στη ζωή τους ε, εκδηλώσεις βίας. Η συζήτηση όμως αυτή έγινε με αφορμή μιας άνευ προηγουμένου επίθεσης στην κολονία. Μιας επίθεσης ε, εις βάρος γυναικών την ε, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, το βράδυ της πρωτοχρονιάς και μάλιστα οι δράστες ήταν ε, κυρίως ε, μετανάστες ή πρόσφυγες. Περιμένουμε συγκεκριμένη συμπεριφορά από τους ανθρώπους αυτούς και δεν μπορούμε να υποτιμούμε τους κινδύνους για την ασφάλεια. Θα πρέπει να λάβουμε επιπλέον μέτρα ασφάλειας και μια τέτοια επίθεση σαν αυτή που έγινε στην κολονία. Μερικές φορές ε, εξοργίζει τον κόσμο η βυσβάρος των μεταναστών ή των προσφύγων αλλά δεν μπορούμε να αποσιωπούμε, να αποκρύπτουμε τέτοια περιστατικά. Όταν έχουμε μεγάλη συγκέντρωση και συγχρονισμό ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικούς ε, πολιτισμικούς ε, κύκλους, είναι φυσιολογικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τόσα πολλά συνέβησαν την παραμονή τη πρωτοφανία στην Κολονία και τα άλλε πόλεις που δεν μπορούσαν να ανταγνωρίσουν ούτε τα ΜΜΕ ούτε η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Αλλά δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε πρόκειται για κάτι το καινούργιο, γιατί δεν είναι χρόνια τώρα και δεκαετίες. Μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έχουν υπερεκπροσώπηση στις ε, ευρωπαϊκές στατιστικές σεξουαλικών και βίων εγκλημάτων. Το μόνο πράγμα που άλλασε ήταν, ήταν τα απόλυτα αριθμητικά είναι αφέλεια το να αγνούμε το πρόβλημα, το να θεωρούμε ότι μπορούμε να βάλουμε αυτούς τους νερούς σε μια τάξη σχολείου και να τους διδάξουμε τι σημαίνει η ισότητα των φίλων ε, και έτσι τους μετατρέψουμε σε καλούς Ευρωπαίους ε, ε, είναι φενάκι. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Εάν φέρει στη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη, η Μέση Ανατολή θα φέρει μαζί και τη μεσανατολική της νοοτροπία. Ε, αυτά που κάνουν δεν τα κάνουν επειδή, νομίζουν ότι δεν είναι κάτι το κακό, επειδή θεωρούν ότι είναι κάτι το καλό. Θέλουν μόνο να μας δείξουν ποιος είναι αυτός ο οποίος κυβερνάει στο δημόσιο χώρο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σόγκορ, ένα λεπτό και τρία το δεύτερα. Ευχαριστώ. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτή η βία των γυναικών είναι αποκλειστικότητα των μεταναστών. Δυστυχώς κάθε χρόνο υπάρχουν πολλέ γυναίκε θύματα αυτών των φαινομένων. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τη υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα, μια στι πέντε γυναίκε είχε παρόμοια εμπειρία στην Ευρώπη. Και πολλέ έχουν αντιμετωπίσει σεξουαλική βία πριν τη συνέντευξή του. Δεν μπορούμε λοιπόν όμω να ανηθούμε ότι ήταν κυρίω σε εκείνη περίπτωση κυρίως πρόσφυγες που όχλησαν σεξουαλικά γυναίκες έξω από το σταθμό της κολονίας. Οι δράστες λοιπόν δημόσια όχρησαν τα θύματα τους με τρόπο ο οποίος δεν αποδεκτός στον δικό μας πολιτισμό. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να εξιστοποιήσει τη σημασία του συμβάντος στην κολονία. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτοί που ήταν δράστες αυτών των γεγονότων να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε άσυλο σε αυτούς που πραγματικά προσπαθούν να ξεφύγουν από τις διώξεις και τον θάνατον και δεν θα πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν σε μια, σε μια συνέχιση της βίας. Το κύριο μάθημα μας εδώ θα είναι ότι ως κοινωνίες υποδοχής θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις νοοτροπίες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο αυτό ώστε να ακολουθήσει τις βασικές ε, ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουίτσα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Με βάση μια έρευνα που έγινε το 2012 στο Λονδίνο, 43% των νέων γυναικών δήλωσαν ότι είχαν υποστεί παρενόχληση την τελευταία χρονιά. Ε, μάλιστα οι έρευνες και ε, μελέτες από τη Γαλλία το 2013 έδειξαν ότι μία στις τέσσερις γυναίκες υπέστησαν ε, κάποια παρενόχληση στο δρόμο ή λεκτική παρενόχληση. Έχουμε λοιπόν τέτοια φαινόμενα εις βάρος γυναικών και παιδιών που αντιμετωπίζουν σε όλους τους κύκλους της ζωής και εμποδίζουν την, την ε, πρόσβασή τους σε κάποιες ε, δραστηριότητες αναψυχής και πειράζουν αρνητικά την υγεία τους. Να δούμε τα επεισόδια της κολονίας. Φυσικά ε, δεν θα πρέπει στην Ενωμένη Ευρώπη να επιτρέπουμε να μην μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα τα κορίτσια, οι γυναίκες μας στους δημόσιους, χώρες, στους δημόσιους χώρους. Πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτά δεν είναι απλά παραπτώματα. Αυτή η συμπεριφορά είναι εγκληματική συμπεριφορά αξιόπινη και θα πρέπει οι δράστες να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο έναντι πάντων. Και δεν θα πρέπει σιλίδιν να καταδικάζουμε τους μετανάστες ή τους ξένους ή τους πρόσφυγες, αλλά να εφαρμόσουμε τον νόμο παντού και σε όλους. Και θα πρέπει να τον εφαρμόσουμε και σε όσους έρχονται στην Ευρώπη από τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε μια θεμελιώδη αρχή και αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Τελευταίος, τελευταία ομιλητρία πριν το Κατστιά, η κυρία Πέτσιρε να λεπτό. Ευχαριστώ. Κάθε διαξίζει κατά δίκης. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ή καμία συνθήκη που να δικαιολογεί τέτοια βία. Δυστυχώ όμω, οι γυναίκε όλο και πιο συχνά γίνονται θύματα βία, ιδιαίτερα σεξουαλική, και πολύ συχνά συζητούμε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα περιστατικά όμω που τελευταία αντιμετώπισαν πρόσφατα πολλέ χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνούν το θέμα τη προστασία των γυναικών και τη καταπολέμηση τη βία βάρο των γυναικών. Τα αποτρόπια αυτά επεισόδια, εκτό από τα θύματα έφεραν στο πρώτο πλάνο και τους δράστες αυτών των φρικτών εγκλημάτων. Δεν θα πρέπει φυσικά να γενικεύουμε και να καταδικάζουμε σιλίδιν όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες για αυτά που συνέβησαν, αλλά δεν θα πρέπει ούτε να παραβλέπουμε ότι ε, οι δράστες δεν ήταν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καθήκον να το κάνουμε. Όχι απέναντι μόνο στις γυναίκες που ήταν θύματα της βίας, αλλά και απέναντι στους πρόσφυγες που προσπάθησαν να γλιτώσουν από τον πόλεμο και να αναζητήσουν προστασία στην Ευρώπη. Γιατί και για τη δική τους ασφάλεια και αξιοπρέπεια θα πρέπει να μεριμνήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται σε αξίες. Πιστεύουμε στην αξιοπρέπεια των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζει τι θεμελιώδει ελευθερίε και τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν δέχεται τη βία ει βάρο των γυναικών σε καμία μορφή. Αυτέ είναι οι πραγματικέ ευρωπαϊκέ αξίε που θα πρέπει να προστατεύσουμε, να προασπίσουμε και να ε, τι ασθενιστούν και όσοι θέλουν να βρουν ένα σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα προσωρινό ή μόνιμο. Ο σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και του νόμου είναι προπόθεση για τη ζωή στην Ευρώπη. Η καταπολέμηση τη βία με την προαγωγή των αξιών μα με την κοινωνική ένταξη και το διαπολιτισμικό διάλογο είναι πράξεις πολύ σημαντικές και σε αυτά θα πρέπει να επενδύσουμε. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Καρσιάη. Τέσσερις συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Η κυρία Ρόχονεν Λέρνα έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. μόνοι στο σκοτάδι. Έτσι βγαίνουν οι γυναίκες στην Φιλανδία για τζόγκινγκ και δεν φοβούνται. Νομίζω λοιπόν εκτιμάμε τις ευρωπαϊκές μας αξίες οι οποίες όμως τώρα δέχονται επίθεση. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να τις προσπιστούμε. Η σεξουαλική ελευθερία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε και να προσπιστούμε τη στιγμή που η σεξουαλικότητα σε πολλά Ισλαμικά κράτη είναι, είναι πρόβλημα και η ομοφιλοφιλία αποτελεί ένα ταμπού. Αυτά οδηγούν δυστυχώς σε συσσόρευση εντάσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα εκραγεί σε άλλα μέρη όπως την κολονία ή το Ελσίνκι. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τις γυναίκες και υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Λίδια Σέντρα Ρούντρικε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η παρενόχληση και η βία βάρος των γυναικών είναι δυστυχώς φαινόμενα σε μια φαλοκρατική αδροκρατούμενη κοινωνία που δυστυχώς δεν ανοίγει τις αγκάλες της ούτε προς άλλους πολιτισμούς, προς άλλες κουλτούρες, ούτε προς τους μετανάστες. Κάθε βέβαια πράξη βίας θα πρέπει να τύχει καταδίκης και τιμωρίας. Πάνω από τις μισές γυναίκες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, νιώθουν φόβο και μερικές φορές αλλάζουν και τι συνήθειέ του για να αποφύγουν συγκεκριμένους χώρους ή καταστάσεις από φόβο μήπω γίνουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης ή βίας. Το 2014, 21 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσαν ότι έγιναν θύματα ε, σεξουαλικής παρενόχλησης από νεαρό ή ε, άνδρα άνω των 15 ετών. 553 δολοφονίες είχαμε στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια. 553 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από φαλοκρατική βία. Μέχρι στιγμή ε, ήδη στην Ισπανία έχουν χάσει τη ζωή του 8 γυναίκε από οικογενειακή βία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Θα πρέπει να αναλάβουμε δραστικά μέτρα και να εφαρμόσουμε συνεπεί πολιτικέ ει βάρο τη φαλοκρατία για την βία πάση μορφή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό κυρία πρόεδρε η σεξουαλική παρενόχληση και η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα χρόνιο κοινωνικό πρόβλημα που εν μέσω οικονομικής κρίσης εντείνεται όλο και περισσότερο. πρόσφατα παρατηρήσαμε τη μαζική σεξουαλική παρενόχληση περίπου 90 γυναικών που έλαβε χώρα στην κολονία για την οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές φαίνεται να είναι υπαίτιοι, αφρικανοί και άραβες την επομένη ημέρα οργανώθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στη βία κατά των γυναικών αλλά και κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της μέρκελ. είναι βέβαιο ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες οφείλουν να ενταχθούν ομαλά στην ευρωπαϊκή κοινωνία για όσο χρονικό διάστημα παραμείνουν προσωρινά στην ευρώπη. ωστόσο η βία κατά των γυναικών είναι ένα πρόβλημα που δεν γνωρίζει εθνικότητα τάξη και κοινωνικά στρώματα ειδικότερα στις χώρες που πλήττονται από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας οι περιπτώσεις βίας σε βάρος των γυναικών καθώς και η ανισότητα των δύο φύλων εντείνεται. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κυρία Γκουστάλ για ένα λεπτό, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μία στι τρει γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί κατά τη ζωή του κάποια φυσική ή σεξουαλική βία. Στην Ισπανία 109 γυναίκε δολοφονήθηκαν από άντρε. Το 2016 μέχρι τώρα έχουμε 11. Πολλές χιλιάδες Γυναίκε νέε είναι αντικείμενο στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν δομικό αυτό το πρόβλημα στην Ευρώπη, τόσο δομικό όσο και το κοινοβουλίο μα. Δεν είναι πρόβλημα άλλων χωρών, το έχουμε στην Ευρώπη. Οι σεξουαλικέ επιθέσει κατά αυτό των Γερμανών γυναικών την παραμονή πρωτοχρονιά αποτελούν θύμα αυτή τη αντίληψη των γυναικών που δυστυχώ διέρχεται όλε τι χώρε, εθνικότητε, πολιτισμού χωρί εξαιρέσει. Το να κάνει κανεί ισλαμοφοβική, ρατσιστική προπαγάνδα αποτελεί ε, μια προσβολή για τα θύματα του, του σεξισμού. Θέλουν λοιπόν να περιορίσουν τις ελευθερίες των γυναικών. Η συνταγή μας λοιπόν κατά του, της φαλοκρατίας και του ρατσισμού είναι η ίδια. Περισσότεροι δημόσιοι υπόροι για μια εκπαίδευση η οποία θα καταπολεμά τα στερεότυπα. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Τώρα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, η κυρία Κόρινα Κρέτσου, Επίτροπος. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για τις προσπάθειές σας να υπογραμμίσετε την ανάγκη να ταθεί ένα τέρμα στη σεξουαλική παλινόχρηση και τη βία εις βάρος γυναικών. Γνωρίζω πολύ καλά τους αγώνες, ο οποίο αποδίδεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων των γυναικών και των εργασιακών βεβαίως, αλλά και στην πολιτική ζωή. Και με λύπη μου αναγκάζομαι να πω ότι έχουμε αρχίσει να μιλούμε για βία. Και δεν ε, μιλάμε, δεν μιλάμε πια για έλλειψη σεβασμού που είναι διάχυτο σε όλα τα κράτη-μέλη. Μιλούμε για βία γιατί δεν μπορούμε να αποστρέψουμε το βλέμμα από αυτό το φαινόμενο ή τα γεγονότα όπως αυτά της κολονίας ή άλλων κρατών, άλλων πόλεων ε, στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα λοιπόν αυτή η συζήτηση για την Ευρώπη και όπως είπα και στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις τα κράτη-μέλη δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας οφείλουν να τεθούν στην πρώτη γραμμή για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της τάξεως. Δική τους είναι η ευθύνη διότι δεν προβλέπεται από τη συνθήκη πουθενά αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θετήσει μια σειρά από νομοθετήματα, ωστόσο, με κοινού κανόνες για την προστασία και την παροχή υποστήριξης σε θύματα εγκλημάτων. Η συναλφός Γιώροβα ασφαλώς θα σας δώσει πιο πολλές λεπτομέρειες στην έρθει ώρα. Υπάρχει ένα εγκάρσιο νομοθέτημα για τα δικαιώματα των θυμάτων εν γέννη. Για τα θύματα βίας ε, φιλετικού χαρακτήρα, μάλλον σεξιστικού χαρακτήρα και για άλλα προστατικά μέτρα. Επίσης εστιαζόμαστε στην υλοποίηση της φυστάμενης νομοθεσίας τώρα, την οδηγία δηλαδή για τα δικαιώματα των θυμάτων. Η Επιτροπή βεβαίως θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί την υλοποίηση, την εφαρμογή από πλευρά των κρατών μελών της φυστάμενης νομοθεσίας πριν προτείνει νέε προτάσεις. Μέχρι τώρα 11 μονοκράτη κράτη-μέλη έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμοστικά τις οδηγίες των οδηγίων μέτρα. Όπως και να έχει θα ήθελα να σας πω πως συμφωνώ μαζί σας στη διαπίστωση ότι πρέπει να καταδικάσουμε αμήλικτα τη βία και να στηρίξουμε τις γυναίκε που έχουν πέσει θύματά της. Η Επιτροπή σκοπεύει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη αξία τη ισότητα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων να καταστούν πραγματικότητα και βίωμα για οποιονδήποτε ζει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Προστασία του. Ε, δεν υπάρχει καμία ε, επιφύλαξη προέλευσης σκεφτικής, εθνοτικής ή ιδιωτικού βίου ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε κανείς να επικολεστεί για να δικαιολογήσει την ε, βία εις βάρος των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση.